Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να κρατήσετε τις θέσεις σας. 19. Ιανουαρίου 2012 διακόπη συνεδρίες, η οποία τώρα συνεχίζεται τα πρακτικά της συνεδρίας της 19ης Ιανουαρίου 2012 και τα εν λόγω κείμενα είναι ενώπιόν σας. Υπάρχουν διαφωνίες, παρατηρήσεις. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά αυτά. Πέραμε σε